So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Herzlich willkommen zu unserer Καλώς ήρθατε. Στη σημερινή μας συνεδρίαση ο ήλιος λάμπει έξω. Δεν, είχε, δεν έχει ποδόσφαιρο σήμερα το πρωί, το απόγευμα έχει. Ε, έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες όμως. Ελπίζω όλοι να έχετε τις κάρτες των ψηφοφοριών σας. Θα τις χρειαστούμε σίγουρα. Und dann äh, Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις ψηφοφορίες για το σημείο 8 ε, της ημερήσιας διάταξης. Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτώνων. Της Κρίστα Κλάς. κλείνουμε τις ε, κουρτίνες για να μην μας τραβώνει ο ήλιος, να βλέπουμε ποιος είναι παρόν. Ποιος σηκώνει το χέρι και ποιος όχι. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις πληροφορίε. Κρίστα, κοίτα αν είμαστε όλοι παρόντες. Ας δούμε πρώτα. Ε, Μήπως τυχόν και έχει κάποια πολιτική ομάδα κάποιο ψήφο παραπάνω. Ε, ας ψηφίσουμε λοιπόν. Ο καιρό είναι ωραίο ή άσχημο σήμερα. Αρχή τη ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Λοιπόν, λειτουργεί το σύστημα. Κανείς δεν ήταν, ε, σχεδόν κανείς δεν ήταν κατά. Λοιπόν. Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Μάλλον όχι. Η πρώτη ψηφοφορία είναι 103 Γιόργενσεν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έχουμε μία ενοποιημένη τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ. Και μάλιστα βλέπω ότι κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ θα ψηφίσουμε ξεχωριστά σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Abstimmung beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. 50 ψήφισαν, 24 υπέρ, 24 κατά, 2 αποχές. Δεύτερο μέρος, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται μου φαίνεται, αλλά να το ελέγξουμε και αυτό. Αρχή της ψηφοφορίας. Abstimmung beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25 υπέρ, 24 κατά. Τρίτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Να το ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην ε, επιτροπολογία ευθυγράμμιση με την συνθήκη της Λισαβόνας της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 1, τροπολογία 10, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 128, σε δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος μόνο. Τις 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήμκο 6. Καταπίπτει. Ήμκο 7. Καταπίπτει επίσης. Επόμενη σελίδα. Ήμκο 8 ως προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 2. Όμοιες είναι 129, 130, Ήτρε 9 και Ήμκο 9. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Und beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, 24 κατά. 131. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δώδεκα υπέρ κατά, αποχές, να ελέγξουμε την δώδεκα. Und Abstimmung beendet. Λήξη Απορρίπτεται. 24 υπέρ, 26 κατά. Άρθρο 3. 13 υπέρ. κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14, ΙΜΚΟ 10, Ήτρε 10, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά αποχές θα έλεγα ότι εγκρίνεται αλλά το ελέγξουμε Beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Ναι, εγκρίνεται με μικρή διαφορά. 134 μότι υπέρ κατά Το ίδιο περίπου, αλλά να ξαναδοκιμάσουμε, να το ξαναλέξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 27 κατά. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 καταπίπτει, 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 καταπίπτει. Προχωράμε στην 139, Κέρπερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 16 και η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Ουί. Απορρίπτεται. Es geht weiter mit 140 Jürgensen. Προχωράμε στην 140 Jürgensen. Jürgensen. Ποιος είναι υπέρ? 140. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. στην επόμενη σελίδα 21 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 141. σαράντα Ποιος είναι υπέρ. 141, 142, ήτρε 17 και ΙΜΚΟ 13. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές να το ελέγξουμε. Beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ήτρα 18, 145, 147, ΙΜΚΟ 14. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ήτρα 19, 145, 148, ΙΜΚΟ 15, υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνονται. 145 μπουσόι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 20, 16, 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 146 καταπίπτει. Επόμενη σελίδα. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 322 καταπίπτει. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29 υπέρ, 27 κατά. Η 144 καταπίπτει. Η 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 4. 150 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε. Abstimmung beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Knapp, aber... Μικρή διαφορά. Εγκρίνεται όμως. Έχουμε όμοιες τροπολογίες, την 151, ήτρα 24 και ΙΜΚΟ 18. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152, 155, παράγραφος 2α. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155, παράγραφος 2β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 καταπίπτει. 25, ή 25, ήμκο 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 26 της εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, μου φαίνεται πως είναι πάλι η δια, ε, διαφορά, αλλά να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας για την 154. beteiligen sich nicht mehr alle. Δεν συμμετέχουν πια όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Καλύψαμε πολλά με τις συμβαστικές τροπολογίες. Μπορούμε να προχωρήσουμε Ja, Seite 14 geht es mit Artikel 6 weiter. Προχωράμε στο άρθρο 6. 14. Σελίδα 14. Also, Sie haben andere Seitenzahlen, sorry. Έχετε άλλες ε, σελίδες. Ε, καλά, σελίδα 14 δική μου είναι. Εν πάμε στο άρθρο 6 με τις όμοιες τροπολογίες 30, ε, Ήτρε 30 και ΙΜΚΟ 23α. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 181 ριβάζει υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όμοιες είναι η 31, η 331, η 23β. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, δεν ψηφίζουν όλοι. Οι φιλελεύθεροι τι ψηφίζουν, δεν είδα. Για πάμε πάλι. Ποιος είναι υπέρ της 182. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. 182. Λήξη της ψηφοφορίας υπέρ. Απορρίπτεται. 183 ριβάζει. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. 183. Λήξη της ψηφοφορίας. εγκρίνεται με μικρή διαφορά. Αλλά δεν ψηφίζουν όλοι πάντα. Μήπως κάποιος ξεχνάει να πατήσει το κουμπί. Εγκρίνεται. 184 ριβάζει υπέρ. Κατά. Θα το ξαναελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Αυτή τη φορά ψήφισε ένας παραπάνω. Η λήξη της ψηφοφορίας ε, και έχει διαφορά το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Ήταν χρήσιμη η, παρατη... Ήταν χρήσιμη η παρατήρησή μου για κάποιους, όχι για άλλους. 185-186 είναι όμοιες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Προχωράμε στην 190 ριβάζι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. So beendet. Λήξη τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Άρθρο 7. Ήμκο 24. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όμοιες είναι η 32, ήμκο 25, ήτρε 32. Ποιος είναι υπέρ? κατά Αποχέ εγκρίνεται. Όμοιε είναι η 33, η ΙΜΚΟ 26, η 33. ποιο είναι υπέρ? Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Η 34 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Όμοιες είναι η 34, η ΙΜΚΟ 27. Ποιος είναι υπέρ? κατά αποχές εγκρίνεται. 35, Ήτρε 35, Ίνκο 28, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 8. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 192 dafür. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193. Κατά αποχές εγκρίνεται. Artikel 9. 31. Κεφάλαιο, ε, άρθρο 9, συγγνώμη, Imco 31, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όμοιες είναι 195-196, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. E το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ναι, ήταν πολύ αποτελεσματική η κινητοποίησή μου, αλλά ωραία, το διορθώσαμε. Απορρίπτεται. 28 υπέρ, 29 κατά. 199 υπέρ. κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία, αλλά ας το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Δύο ψήφοι λείπουν. Αλλά αν δεν πατήσετε το κουμπί, Λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αλλά δεν ψηφίζετε όλοι. Οι επόμενες καταπίπτουν. Προχωράμε στην 200. 201 ΙΜΚΟ 31 Β με χωριστή ψηφοφορία σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. «202. Μέρκης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 203, 204, 205 είναι όμοιες. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. ended. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31 υπέρ, 26 κατά. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε. 206. Το ΕΛΚ έχει μία ψήφο παραπάνω. Κύριε Ούλμαν, ευχαριστώ. Θα πρέπει να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Η 29 υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται. Καλύτερα να ψηφίζουν αυτοί που έχουν κάρτα, διότι λείπουν τρεις που δεν ψηφίζουν αλλά είναι παρόντες. 207 προχωράμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 31 δέλτα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Γίτσες. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 211 ή 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έχει αποσυρθεί η 2.13, οπότε προχωράμε στην 2.14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μικρή διαφορά. Νομίζω εγκρίνεται. Άλλωστε ελέγξουμε. 2.14 ψηφίζουμε. Λήξη. Εγκρίνεται. Άρθρο 10. 2.16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 2.18. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Άρθρο 11. Ή 340 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προχωράμε στο άρθρο 13. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.22 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ε, Ήτρε 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 15. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 229, 230, ΙΜΚΟ 34, 228, ΙΤΡΕ 43. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 40.41, σαράντα ΙΜΚΟ 35, Ήτρε 44, 45. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όμοιες είναι 2.31, 2.32 ή 3.46, ΙΜΚΟ 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται, θα το ελέγξουμε. 233. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 234. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε. 234. Λάθος είδα. Εγκρίνεται με σημαντική διαφορά. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λάθος μου. Ωραία, άρθρο 16. 235 της κυρίας Βίλς. Ποιος είναι υπέρ. 235 της κυρίας Βίλς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 238 καταπίπτει. Η 239 καταπίπτει. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 ή 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 243 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 244 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 45, ΙΜΚΟ 38, Ήτρε 49. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 39, Ήτρε 49, 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 246 υπέρ κατά άποχέ εγκρίνεται. 247 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 248 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όμοιε είναι οι 47 και οι 350 χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 ή 51 ή 40. ε, συγγνώμη, ή 51. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 40 υπέρ επακαταπίπτει. Άρθρο 17. 249 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 250 ή 352. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 52. Παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1, υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Ήτρε 52, σημείο Β, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 251, ποιος είναι υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 52. Σημείο Γ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 52. Εισαγωγή. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιώργενσεν 254 χωριστή ψηφοφορία σε τρία μέρη. Πρώτο μέρος ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε το τρίτο μέρος. Το ΕΛΚ έχει μια ψήφο παραπάνω. Μια κάρτα πρέπει να βγάλετε. Τώρα είμαστε εντάξει. Δύο έβγαλαν τι κάρτε του. Τέλος, πάντων του ή καμία διαφορά απορρίπτεται. Και φτάνουμε στην 255 υπέρ. Πλουμ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 352 β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 257. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές απορρίφθεται. 258 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, 258 να ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ναι, όπως είπα, εγκρίνεται. Έτσι είναι. Η 352 καταπίπτει. 259 Wills υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 260, 261 είναι όμοιες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 265 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 264 το σημείο CA υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 264 το σημείο CB. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 264 σημείο CC υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 268-269 ή 352. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Imco Wer ist dafür? Ήτρε 52. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 18. 49 Ήτρε 53 υπέρ. Καταπίπτει. επειδή απορρίψαμε την 16 πίπτη. Η 50 καλύπτεται από συμβασική τροπολογία. 273 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 274 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 51. Το υπόλοιπο του κειμένου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52. Ήτρε 54 καταπίπτουν. Πενήντα τρία. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όμοιες είναι 2,75, ΙΜΚΟ 42, καταπίπτουν. 54 είναι η επόμενη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 19, 276 Γιώργενσεν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 277 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 20. Ψηφίσουμε την 55 ή 57 ή 44 που είναι όμοιες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. «280 Γιόρκενσεν υπέρ». Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρα 59 υπέρ. Κατά αποχε εγκρίνεται. 282, 283, 284, Ήμκο, 46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Ήτρε 60, καταπίπτει. Ήτρε 61, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Όμοιες είναι 285, 281, ΙΜΚΟ 47. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 21. Όμοιες είναι 286, 288, Ήτρε 62. Χωριστή ψηφοφορία, το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την ΙΜΚΟ 48. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Η 289 αποσύρεται. Ήτρε 63, ΙΜΚΟ 50, 292, 311. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 290. Καταπίπτει. Ητρε über 65. ITRE α. Είναι η επόμενη που θα ψηφίσουμε. Ητρε 65 σε μία α. Ποιος είναι υπέρ? Dagegen. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ein Μία ψήφο παραπάνω έχουμε από το ΕΛΚ. Ωραία, τώρα εντάξει. Λήξη της ψηφοφορία. εγκρίνεται. 31 υπέρ. 27 κατά. Όμοιες είναι οι 296, 298. Ποιος είναι υπέρ? Ακαταπίπτουν. 300 είναι η επόμενη. Ήτρε 65, 301. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 302 μόνο το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην 303. Όμοια με την 304. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. 303 και 304 που είναι όμοιες κατά. Αποχές απορρίπτονται. 306 έχει αποσύρθει. 308 είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 309 Κράμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 310 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 22. Όμοιες είναι 57 έως 61 και ήτρε 67. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Λοιπόν, να ελέγξουμε την προηγούμενη ψηφοφορία. 57 61, ήτρε 67. Εγώ είπα ότι εγκρίθηκα, να το ελέγξουμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Όλοι είναι υπέρ. 49 υπέρ, 9 κατά. Ίσως να ήταν λάθος στη μετάφραση. Άρθρο 23. 312 ή 368 ήμκο 60. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όμοιες είναι 62 ή 69. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. Ήτρε 72. 70, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Dann Artikel 24, identisch. Άρθρο 24, όμοιες είναι η 313, ήτρε 71, η 61. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 25. Ήτρε 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Abstimmung beendet. Angenommen. Εγκρίνεται. Ωραία. Όμοιες είναι η 275, η 42. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 62-63 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όμοιες. Μάλλον καταπίπτουν. 315. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 27. Όμοιες είναι η 316, η 375, 76, η ΙΜΚΟ 64, 65. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 28. Όμοιες είναι η 317, η 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.17 πίπτη. Ή 3.77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 67. Ναι, υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. Λήξη. Εγκρίνεται. Υπάρχουν κάποιοι που δεν σηκώνουν κάτω το χέρι τους και είναι δύσκολο να δει κανεί. Λοιπόν, έχουμε όμοια στην ΙΜΚΟ 68 και 318. Ποιος είναι υπέρ? Καταπίπτει. Ήτρε 78. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές Αποχή Άρθρο 29. 319 ριβάζει. Ποιος είναι υπέρ? κατά, αποχές, να το ελέγξουμε. 3.19. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά. 3.20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. 3-20, αρχή της ψηφοφορίας. Κάριν, να βγάλεις την κάρτα σου. έχουμε μία ψήφο παραπάνω. Ή κάποιος άλλος. Ωραία, τώρα είμαστε εντάξει. Εγκρίνεται. 321. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε και πάλι. 321. Κυρία Κορτίνες, δεν είναι απαραίτητο. Έχουμε μια ψήφο παραπάνω. Μπορείτε να βγάλετε την κάρτα σας. Ωραία. Εγκρίνεται. 322 Μέρκης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 323 Μέρκης. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 324. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 325 που είναι όμοια με την Ήτρε 79 και την Ήμκο 70. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όμοιες είναι η 326, η 380, Ήμκο 71. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 31. 328 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 329. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 327 ριβάζει. Ποιος είναι υπέρ. Όχι, θα την ψηφίσουμε ότι καταπίπτει μόνο εάν απορριφθεί η 328. Ψηφίσουμε λοιπόν την 327. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές να το ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Da der dritte Teil des konsolidierten Änderungsantrages abgelehnt το τρίτο μέρος της ενοποιημένης ε, τροπολογίας ε, απορρίφθηκε, γι' αυτό πρέπει να τις ψηφίσουμε αυτές, γιατί δεν καταπίπτουν. Yeah. Hm. Dann geht's los mit Itra 1. Πάμε λοιπόν, Ήτρε 81, παράγραφος 1, α, 1. Ε, ποιος είναι υπέρ? Ήτρε 81, παράγραφος α, λέει ο Πρόεδρος. Κατά. Να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται. So, es geht weiter bei 331. Προχωράμε με την 331 ριβάζει. Ποιο είναι υπέρ τη 331. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 331. Abstimmung beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 64, 339, 340, 341, 342. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 Also ich höre, wir stimmen über IMCO 73 ab. IMCO 73 ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ. Άρθρο 33α. Ποιος είναι κατά τη ΣΥΜΚΟ 73. Να το ελέγξουμε. Ο Χόλκερ Κράμερ με ενοχλεί. Διότι ψηφίζει πάντα το αντίθετο από του υπόλοιπου φιλελεύθερου. Αυτό με ενοχλεί. Μα αποφάσισε επιτέλους με ποια πλευρά είσαι. Εντάξει, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ωραία. Άρθρο 34, όμοιες είναι οι 65 και οι 82. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. μικρή διαφορά, ας το ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Άρθρο 35, όμοιες είναι 66 ή 383. Ή αυτές οι δύο. Ποιος είναι υπέρ. κατά, αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 84. Ήτρε Ποιος είναι υπέρ, Ήτρε 84 κατά, αποχές απορρίπτεται. 67 της εισηγήτριας, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 3.46 ή 3.85 ή 74. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.47 Γιώργενσεν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.48 Γιώργενσεν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 351 ήτρε 86. Ποιο είναι υπέρ της 351 και της ήτρε 86. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 352. Καταπίπτει. Άρθρο 36. Όμοιες είναι 353, 354 ή 387 ή ΙΜΚΟ 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 37 ή 388 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 37α. Τι πρέπει να εδώ. Προχωράμε, άρθρο 38, 355, ρίς λεπάς, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όμοιες είναι η 70, η 91, η 76. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 39, 356, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 357, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 40. Το πρώτο μέρος μόνο. 71 της εισηγήτριας, ή 93 το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 41. 41 haben wir nichts abzustimmen, weil alles wegfällt. Στο άρθρο 41 δεν ψηφίζουμε τίποτα γιατί όλα καταπίπτουν. Άρθρο 42 το κοιτάμε ένα λεπτό. Εβδομήντα ψηφίζουμε. Στο άρθρο 42 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 96 dafür. υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Α, άσχημα τα πράγματα κυρία Κλάση. Dann 362, 363. 362, 363, 78. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 44. Έχουμε πολλές όμοιες, από την 365 μέχρι την Ήτρε 98 το πρώτο μέρος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όμοιες είναι 368, 369, Ήτρε 98, ποιος είναι υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται. «370», «ΙΜΚΟ 80», «ΙΤΡΕ 98», ποιος είναι υπέρ. Κατά, άποχες εγκρίνεται. Όμοιες είναι η 371, η 80, η 398, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρακόσια εβδομήντα τέσσερα, ΙΜΚΟ ογδόντα, ΙΜΚΟ 98, λέει ο πρόεδρος, ή ημάνου, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 99 και Ήμκο 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 375 Ήτρε 100 Ήμκο 82. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 45. 376. 378. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 46. Ήτρε 101 υπό παράγραφος 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε 379 έως ήτρα 102 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Τρία ογδόντα μότι, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, να το ελέγξουμε. Μότι 380 αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αυτό είπα. Ήμκο 83. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτουν όλες οι επόμενες 3. 86 Σουλή Κροστέτ Φράγκο είναι όμοια με την 387, 388, ΙΜΚΟ 83. Ποιος είναι υπέρ. Δεν έχει αγγλική μετάφραση, τι κρίμα. Ακούτε τώρα. Πάμε πάλι 386 έως ΙΜΚΟ 83. Είναι το μπλοκ που ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Λείπουν τέσσερις που θα μπορούσαν να ψηφίσουν. Λήξη της ψηφοφορίας όμως. Εγκρίνεται. 3, 89, ΙΜΚΟ 83, ΙΤΡΑ 103. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα πρέπει να ελέγξουμε Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Απορρίπτεται. 390 μότι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 391 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 47. 393 Weisgerber υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. 393 επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. 394 μπούζο υπέρ. Κατά. Ε, κουραζόμαστε, βλέπω, οπότε η ηλεκτρονική επαλήθευση 394 μπουζού. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. 395 ε, γκίρλινγκ υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 396 ντελάγγι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 414 πυρίλα και ήτρε 106 414 πυρίλο και ήτρε 106 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Κατόπιν ΙΜΚΟ 84 υπέρ. ΙΜΚΟ 84 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ταυτόσημες η 397, 399 και η 104 με προφορική τροπολογία και χωρίς την ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μετά 398. Ριβάζει υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τετρακόσια τέσσερα, με την 405, Μπουζόη και Πυρίλο, υπέρ. κατά αποχές εγκρίνονται. Ταυτόσημες 77, 408 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 407 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε στην Ήτρα 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Για την Ήτρα 105. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται. 412 Βάις Γκέρμπερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 84 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 48 ταυτόσημες η 79, η 307 η 85, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ταυτόσημες η 80, η 308 η 86, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ταυτόσημες η 81, η 309 η 87, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άρθρο 49. Ίμκο 88, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όμοιε είναι οι 84, ΕΜΚΟ 88 ή 310 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Όμοιε οι 85, ΕΜΚΟ 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 50. Έχουν αποσυρθεί αυτές. 51, 417 μότι υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Und beendet. Λήξη. Εγκρίνεται 30 υπέρ 28 κατά. 87 της εισηγήτριας ή 311 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 52, 418, Βάισκερπερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 88. Έτσι η αλλαγή. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ήμκο 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 53. Άρθρο 53. Όμοιες είναι 89, Ήτρα 112, Ήμκο 91. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 54. Ήμκο 92 και 90 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 420 είκοσι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 93 καταπίπτει. 421 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 422 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4.23 λεπάζ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4.24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.25 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται Άρθρο 55, όμοιες είναι 426 ή 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 427 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ομοια είναι 428, ΙΜΚΟ 97, ΙΤΡΑ 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ομοια είναι 428, ΙΜΚΟ 98, ΙΤΡΑ 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Όμοιες είναι 428, ΙΜΚΟ 99, ΙΤΡΕ 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Λήξη. Εγκρίνεται. Όμοιες είναι 428 ΙΜΚΟ 100 ή 314. Σημείο DD. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 4.29 λεπάζει υπέρ. Εγκίγν. κατά αποχές εγκρίνεται. 92 ή 315 υπέρ. Dagegen. Enthaltungen angenommen. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 56, 4.30 τα πάτζι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4.31 υπέρ, κατά αποχές Η κυρία Κλάσελη, ε, να το ελέγξουμε, να το κάνουμε λοιπόν κατευθείαν. Λήξη. Εγκρίνεται. 4.32 Μέρκης υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 Ήτρα 116 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. 93 και ήτρα 116. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 4.33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 57. 4.34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 58. Όμοιες είναι 436, ΙΜΚΟ 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 437 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 438 χωριστή ψηφορία, πρώτο μέρος υπέρ. κατά Να το ελέγξουμε. 4.38 το πρώτο μέρος. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. κατά Να το ελέγξουμε το δεύτερο μέρος. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τέσσερα τριάντα υπέρ. κατά, αποχε εγκρίνεται. Όμοιε είναι 440 ή 317 υπέρ, κατά, Κατά, απορρίπτεται. Ήμκο 102 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται. 441 ρίς λεπάς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 442 καταπίπτει. 443 λεπάζει υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 103. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 59. Ήμκο 104. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 61, 94 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 62, όμοιες είναι 445 και ΙΜΚΟ 105 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 446 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Άρθρο 65. Καταπίπτει. Άρθρο 66, ήτρε 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4,48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 70. Όμοιες είναι 4,49, 4,50, ήτρε 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 451 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όμοιε είναι 95 4.52. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Βάις Κέρπερ 456 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 73 Θα πρέπει να ψηφίσουμε την 455, Ροτ Μπέρεντ, μου λένε. Ποιο είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η κυρία Κλάς αγαπάει τους ελέγχους να το ελέγξουμε. Λοιπόν, 455. Abstimmung, ja, beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Ε, απορρίπτεται. Άρθρο 73, 462 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 75-123. Ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 76. 464 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 464. Αρχή της ψηφοφορίας. Ελέγχουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 465 dafür. 465, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 466 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 77. Όμοιες είναι 470, ήμκο 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όμοιες είναι η 96, ήτρα 124, ήμκο 108 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όμοιε είναι 471, έμκο 109, συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 80, 97, υπέρ. Κύριε Ρώση, θέλετε κάτι να πείτε, έχετε διαδικαστικό. Ήθελα να πω όπως ότι υπάρχει κάποιο μικρό πρόβλημα στο ρυθμό που ακούω την, την διαρμηνία και δεν μπορώ να παρακολουθήσω ακριβώς τι γίνεται. Okay. Να τα λέω πιο αργά δηλαδή. Δεν ξέρω, ίσως ε, να μην είναι, να μην είναι ο δικός σας ρυθμός, είναι ο ρυθμός του διερμηνέα. Λοιπόν, 97 ε, της εισηγήτριας, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 81. 472 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 473 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 473 την ελέγχουμε. Λήξη. Τη ψηφοφορία απορρίπτεται. 474 ε. ΙΜΚΟ 111. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 82. Όμοιες είναι 475, 476, Ήτρα 125, Ήμκο 112. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Μικρή διαφορά, αλλά πράγματι απορρίπτεται. Φτάνουμε στα παραρτήματα. Η κυρία Κλάσκα θέλει να πει. Παρακαλώ. Ναι, φτάνουμε στα παραρτήματα. Υπάρχουν πολλές τροπολογίες που είναι κατά των ε, πειραμάτων σε ζώα. Είμαι και εγώ υπέρ του να μην κάνουμε δοκιμές σε ζώα ή ε, ε, να τι περιορίσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν. Επί τη αρχή λοιπόν θα συμφωνούσα με τι τροπολογίε αυτέ, αλλά χθε έκανα κάποιε έρευνε και υπάρχουν κάποιε αντιφάσει. Από τη μία μεριά ζητάμε ελέγχου και πιο αυστηρά κριτήρια, από την άλλη δεν θέλουμε να στηρίξουμε την έρευνα. Μου είπαν ότι όσον αφορά ε, την κληρονομικότητα θα πρέπει να γίνουν περισσότεροι, ε, περισσότερες δοκιμές όσον αφορά τις ε, ουσίες που βλάπτουν το ενδοκρινικό, το ε, ανοσοποιητικό. Ε, κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν μπορώ να εκτιμήσω τι περιλαμβάνεται σε αυτές τις ε, τροπολογίες. Θα ήθελα όμως να προτείνω σήμερα να τις υπερψηφίσουμε, να το εξετάσουμε αυτό, να το ξανασκεφτούμε. Εάν λοιπόν η Επιτροπή μας ψηφίσει υπέρ των τροπολογιών αυτών, θα προκαλέσουμε έτσι περαιτέρω συλλογισμό για το θέμα αυτό και θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Κομισιόν πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για να ξέρουμε τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτές τις μεμονωμένες ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Αν κατάλαβα σωστά, ε, θεωρείτε ότι είναι σωστό να κάνουμε ε, ψηφοφορία on block, να ψηφίσουμε όλες μαζί τις ε, τροπολογίες. Ε, και να ζητήσουμε από την Κομισιόν να εξετάσει αν υπάρχουν αντιφάσεις ε, στα σημεία αυτά. Ε, κυρία Χάση. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, αλλά δεν συμφωνώ με αυτή την ε, συνολική ψηφοφορία για το παράρτημα 2. Η ομάδα μου ζητάει μια ξεχωριστή ψηφοφορία για το 479 και το 480 συν 500, 504, 7, 8, 9 και 10, 516, 528, 530, 33 και 52. Και η Προεδρία έχει ούτως ή άλλως τον ίδιο κατάλογο. Good. Ich habe die Anmeldung bekommen. Also wir haben, Äh Ωραία. 14 από 73 αυτά που είπε η κυρία Χάση. Ε, να ψηφίσουμε ξεχωριστά αυτές τις τροπολογίες. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 73 14 είναι σχεδόν 60 τροπολογίες που θα ψηφιστούν unblock. Προτείνω λοιπόν να τις ψηφίσουμε αυτές μεμονωμένα. Λοιπόν, μπορούμε να ψηφίσουμε το μπλοκ χωρίς αυτές που αναφέραμε, τις έχω σημειώσει. Ψηφίζουμε λοιπόν unblock, μπλοκ, ε, εκτός από τις τροπολίες που ανέφερε η κυρία Χάση. 477 παράτημα 1. Ποιος είναι υπέρ. 477 παράρτημα 1 ριβάζει. Ποιο είναι υπέρ, άλλη μια φορά για να σα δω, κατά. Θα πρέπει να το ελέγξουμε αυτό. Ελέγχουμε 477. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 4,78 ριβάζει ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4,79 και 4,80 πρώτα ξεχωριστά, γιατί αυτό ζητήθηκε. Ποιος είναι υπέρ, τις ψηφίζουμε μαζί αυτές, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Να το ελέγξουμε αυτό. 4,79, 4,80 να τις ελέγξουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το μπλοκ μέχρι την 499 από την 481 έως την 499. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Με μονομένες ψηφοφορίες τώρα το 50, ποιος, 500, ε, συγγνώμη, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 501. Να ελέγξουμε την 500. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 501. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μου φαίνεται ότι έχουμε την ίδια πλειοψηφία. Μου φαίνεται ότι και αυτή απορρίπτεται. Να το ελέγξουμε. Λήξη της συνεδρίασης. Πολύ ενδιαφέρον. Εγκρίνεται. Ε, Πηδάμε τώρα λίγο, θα ψηφίσουμε αυτές που είπε η κυρία Χάση. Προχωράμε λοιπόν στην 504 για την οποία ζητήθηκε ξεχωριστή ψηφοφορία. 504 λοιπόν. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. 504. beendet. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 507. Ποιος είναι υπέρ. Κέρλινγκ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. beendet. Angenommen. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 508. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 509. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται, αλλά μήπως θα το ελέγξουμε. Όχι, εγκρίνεται, 509. 510 υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5-16 είναι η επόμενη που ψηφίζουμε ξεχωριστά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5-28, πηδάω λίγο, Γιώργενσεν, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ε, υπέρ, 528, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 530 Γιούργενσεν. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 533 Γιούργενσεν. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Και ακόμα 5.52. Γκέρλινγκ. 552 πενήντα Γκέρλινγκ. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Και αυτή εγκρίνεται. Λοιπόν, Ψηφίζουμε τώρα σε μπλοκ όλες τις υπόλοιπες που δεν ψηφίσαμε ξεχωριστά. Ποιος είναι υπέρ των υπόλοιπων τροπολογιών on block. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Αυτό μας διευκολύνει αρκετά. Έχουμε κάποιε ε, τροπολογίες που δεν περιλαμβάνονταν στον μπλοκ αυτό. Θα πρέπει να τις ξανακοιτάξουμε. 511 ριβάζει. Τις ε, βρήκατε ποιο είναι υπέρ τη 511. Είναι διαφορετικές οι σελίδες, είναι διαφορετική η αρρύθμιση Στι δικέ μου σελίδε από τις δικές σας. Ε, σε μένα είναι σελίδα 56. Εν πάση περιπτώσει 511 ποιο είναι υπέρ κατά. αποχέ. εγκρίνεται. Έχουμε από το παράρτημα 3 την τροπολογία 100 της εισηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 531 ριβάζει. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 και ήτρα 129 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5.35 και ΙΜΚΟ 116 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Φτάνουμε στο παράθυμα 4. 554 Wheels υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 555 υπέρ, κατά, αποχές. 556 με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνονται ομοιε είναι 5,57, 5,58 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 5,59, 5,60. Είναι γλωσσικέ αυτές μόνο. Δεν χρειάζεται να τι ψηφίσουμε. 5,61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 562 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράδειγμα 5. 563 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Όμοιες είναι 564, 565, 566, Ήτρα 130, Ήμκο 117. Ποιος είναι υπέρ? κατά, αποχές απορρίπτονται. Παράρτημα 6. 567 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Beendet ist angenommen. Εγκρίνεται. 568. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Το ίδιο, νομίζω το ελέγξουμε, 568. Ja, ναι. noch jemand? Άλλος. Dann ist die Abstimmung beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Και εδώ μικρή διαφορά. Ωραία. Λέει εδώ voting block, να τις ψηφίσουμε μαζί, 569, 570, 571, 572, υπέρ. Κατά. αποχές, να το ελέγξουμε. Will noch einer? Ja, kam noch einer. Άλλος? Α, είχαμε άλλον έναν. Εγκρίνεται λοιπόν. Λήξη της ψηφοφορίας. 5.73, ριβάζει. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 574 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 175 λέει ο πρόεδρος, 575 μάλλον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 576 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. 576. Ja, alle abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. 577. Ριβάζει υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 578 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 579 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 580 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φτάσαμε στα εκτιμώντα 104 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται prüfen mal gerade, was noch abgestimmt werden muss und was nicht. Okay. The vote on 109, the reference to seven years. 109, Rivasi. 109, Ριβάζη. Ε, αναφορά στα 7 χρόνια. Πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ 109. Dagegen. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Dann 110 zurückgezogen. Έχει αποσυρθεί εν μέρη. Bald haben wir es geschafft. Κοντεύουμε, κοντεύουμε. Äh, e Τροπολογία 3 και ήτρε 2. Ε, 112, 113, 114. Ποιος είναι υπέρ? Όχι, δεν καταπίπτει, διότι το τρίτο μέρος απορρίφθηκε της ε, ενοποιημένης τροπολογίες. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 3 που είναι όμοια με την Ήτρε 2. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται. 116. δεκαέξι. Wills, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχέσαι. Ε, εγκρίνεται. 116, να το ελέγξουμε. Abstimmung beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ήτρε 3. Ήτρε 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118, 119 ή 34 ΙΜΚΟ 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. 5, Ήμκο 4, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5, Ήτρε 6, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 και ήτρε 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 127 Ήτρε 8 και ΙΜΚΟ 5 τελευταία ψηφοφορία ποιος είναι υπέρ κατά ε, να το ελέγξουμε Λήξη της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Über Ψηφίζουμε την έκθεση ηλεκτρονικά. ποιο είναι υπέρ. Abstimmung ist beendet. Λήξη της ψηφοφορίας. 48 υπέρ, 5 κατά, 6 αποχές. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Αρχή της ψηφοφορίας. Ja. Wer will noch? Niemand mehr? Ποιο άλλο θέλει, κανένας άλλος. Λήξη της ψηφοφορία. 47 υπέρ, 5 κατά, 6 αποχές. Θερμά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια Κρίστα Κλάς. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά. Ευχαριστούμε όλους που ψήφισαν μαζί μας ε, με τόσο θάρρος ε, και η κυρία Λεπάς θα μας πει τι ανακαλύψαν. Υπάρχουν κάποιες ασυνέφειες, Θα πρέπει να το δούμε και να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ελέγξει πάλι το αποτέλεσμα. Στη δεύτερη ανάγνωση θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Μαραθώνιος ήτανε. Πρέπει ακόμα να ψηφίσουμε τις καταστροφές. Ε, μισή καταστροφή ήταν αυτή η έκθεση, αλλά τώρα έχουμε άλλη μία. Ευχαριστώ τη Γραμματεία για τη βοήθειά της στη δύσκολη αυτή ψηφοφορία, στον πολύπλοκο αυτό κατάλογο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 Πήραμε μια ανάσα να προχωρήσουμε λοιπόν τώρα με την ε, έκθεση του Ζωάου Φερέιρα. Κοινοτική προσέγγιση στην ε, πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Έχουμε μια σειρά ενοποιημένων τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών. Πάμε λοιπόν. C1 του εισηγητή. Ποιο ε, είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. C11. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. C2 υπέρ. κατά αποχές ενγκρίνεται. C19 υπέρ κατά αποχές Συ C10 υπέρ κατά αποχές Συ C3 υπέρ κατά αποχές Συ C7 υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε. Στην C7 ελέγχουμε. Ναι. Also wir haben 53 da. 53 παρόντες. 40 ψήφισαν. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορία εγκρινεται εγκρίνεται. C4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συ 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρινεται συ C6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρινεται συ C21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρινεται συ C8 υπέρ. Κατά. Αποχές Συ C9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. C12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. C14 υπέρ, Συ εγκρίνεται. C17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. C18 υπέρ, κατά, αποχές Συ 17 υπερ κατα αποχες εγκρινεται Συ 18 υπερ κατα αποχες εγκρινεται λιμπε 17 υπερ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Παπαδοπούλου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πώς ψηφίζει το ΕΛΚ. Τι ψηφίζουμε. Υπέρ. Εγκρίνεται τότε. Λίμπε 11, δεν την ψηφίζουμε αυτήν. Ρέγγι 2, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άκρη 11 καταπίπτει. 71 κουτιέρες, κορτίνες και πρόντι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. es weiter mit Liebe 2. Wer ist dafür? Liebe 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Πάμε στη διασυνορική συνεργασία 15 Παπαδοπούλου υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Άκρη 17. Αγκρί 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 Παπαδοπούλου με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λίμπε 12 υπέρ. Κατά Αποχέ εγκρίνεται. Ε, απορρίπτεται. Ε, Άγκρι 34 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 37 Ζήπερα αποσύρεται, άρα πάμε στην 38 ε, Αντωνέσκου Νικολέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ανισότητα αλληλεγγύη με τις περιφέρειες. Ρέγγι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Es geht weiter. Και τώρα πάμε στην Ελίμπε 20 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Λίμπε 20, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ρέγγι 9, επέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 τρεμόπουλος υπέρ, κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται η επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίνεται όντως. Από το support 34 κόρτα Ρώση. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, άγκρι 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περέλο, 45 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 και άγκρι 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 55 Περέλο Ροντρίγκες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 Τρεμόπουλος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αγκρή 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Άκρη 18 υπέρ 28 συγγνώμη κατά αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στην 69 του εισηγητή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 Τρεμόπουλος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Λίμπε 16. Ähm, beendet. Hey, knapp. Also. Μικρή διαφορά εγκρίνεται η Λίβε 16. 70. Αντωνέσκου Νικολέσκου. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1. Παπαδοπούλου. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2. Εστρέλα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3. Εστρέλα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 τρεμόπουλος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπερέρολοτρίκες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 Παπαδοπούλου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 Περέλο Ροτρίκες υπέρ κατά